κατάσταση στη Σρι Λάνκα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους συντάκτες των ψηφισμάτων. Πρώτα ο συνάδελφος Σλούτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι τόσο συχνό να ερχόμαστε εδώ και να χαιρόμαστε για τη λήξη ενός πολέμου, όπως ε, πραγματικά συνέβη το 2009 στη Σρι Λάγκα. Στη συνέχεια συστήθηκε το 2010 Επιτροπή Συμφιλίωσης και έχει αρχίσει και ε, στο μεταξύ η αποναρκοθέτηση. Τον Αύγουστο συστήθηκε μια ερευνητική επιτροπή για ε, τους αγνοουμένους και έγιναν στο μεταξύ στη Βόρεια Επαρχία εκλογές. Όλα αυτά είναι θετικές εξελίξεις. Δυστυχώς υπάρχουν όμως και πάλι μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα διότι Ταυτόχρονα βλέπουμε να έρχονται συγκρούσεις, να γίνονται επιθέσεις σεξουαλικές, ε, απειλές γενικότερα να ε, εκτοξεύονται κατά της ε, δικαιοσύνης και συνολικά υπάρχουν και οι απροστάτευτες χείρες ε, πολέμου, οι οποίες υφίστανται ιδιαίτερες απειλές. Γι' αυτό η Σιλάνκα θα πρέπει αμέσως να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται μια επιτροπή που να εξασφαλίζει ότι εκείνοι που ε, έχουν ε, κάνει εγκλήματα πολέμου, εκατέρωθεν των αντιμαχωμένων πλευρών, να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για να επέλθει και η τιμωρία τους κατατέθηκε μια έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη πράγμα απαραίτητο, αλλιώ θα συστήσει ιδιαίτερη εξεταστική επιτροπή ο ΟΗΕ. Ε, θα πρέπει οι εκκληματίε πολέμου να λογοδοτούν πάντα ενώπιον των δικαστηρίων. Και όταν κάποιος έχει πέσει θύμα ε, βίας, είναι πιο εύκολο να ε, το ξεχάσει, να το συγχωρέσει και να συνεχίσει τη ζωή του όταν βλέπει τον θήτη του και τον δράστη να τιμωρείται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σλίτερ. Η κυρία Γκόμας για ένα λεπτό. Ήδη πολλέ φορέ το Κοινοβούλιο έχει οθετήσει πολλά ψηφίσματα για την κατάσταση της Σρι Λάγκα, τονίζοντας τα προβλήματα στη διαδικασία εθνική συμφιλίωση. Ε, και το 2011 επισκέφθηκε μια αντιπροσωπεία δική μα στη Σρι Λάγκα. Υπήρχαν αμφιβολίε, αλλά θεωρούσαμε ότι η Επιτροπή Συμφιλίωση που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση για να διερευνήσει εγκλήματα πολέμου θα λειτουργούσε. Δυστυχώ, φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει σήμερα. Οι διεθνείς ε, απαιτήσει, προποθέσει, δεν τίθεται σε εφαρμογή, δεν υπάρχει τιμωρία ε, για του υπεύθυνου των εγκλημάτων ε, και η κυβέρνηση επιλέγει να κατηγορεί όσους ασκούν κριτική και ανήκουν σε ανεξάρτητες επιτροπές και υποσκάπτει την δημοκρατία στη Σρι Λάγκα. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο ζητά από την κυβέρνηση να υποστηρίξει τις συστάσεις της κυρίας Νάβη Πιλάη από τον ΟΗΕ ε, και να δημιουργηθεί ένας διεθνής μηχανισμός ανεξάρτητος που θα κάνει μία ουσιαστική έρευνα η συμφιλίωση θα πρέπει να βασίζεται στη δικαιοσύνη. Δίχως αυτή δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες, ο συνάδελφο Βανόρντε. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λίσεκα ε, που μου έδωσε τη δυνατότητα πριν να μιλήσω. Ιδίω ε, ε, κάποιοι από τη διασπορά ε, που δεν έχουν ευχαριστηθεί με την ε, κατάθεση των όπλων από την ε, οργάνωση των Τίγρεων. Ε, τώρα όμως πρέπει να δουν μπροστά. Πρέπει να ξεπεραστούν οι ε, διχάσμοι του παρελθόντος και τα λάθη να μην επαναληφθούν. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ευημερούσα οικονομία και ένα μέλλον για όλους, ανεξαρτήτως εθνικής θρησκευτική προέλευσης. Η κυβέρνηση και οι αρχές του Σρι έχουν κάνει πολλά και τους συγχαίρουμε γι' αυτό, αλλά πρέπει να κάνουν και άλλα. Ε, χάσαμε τον Νέλσον Μαντέλα που έχει αναγορευτεί σε ήρα διότι μετά από πάρα πολλά χρόνια φυλακής χωρίς πικρία ε, πρόβαλε και έκανε πράξη την ε, αρχή της συμφιλίωσης. Δεν θα κάνουμε κηρύγματα εμείς αλλά θέλουμε να κάνουν αυτό το βήμα και ε, στη Σρι Λάνκα, η ε, λογική Ταμίλ ε, να Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Φανόρτεν, ο κύριος Μέρφη για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να μην Ακούμε αυτά που λέει η δεξιά. Δεν φταίνε οι Ταμίλ ε, για τα όσα συμβαίνουν στη Σρι Λάνκα. Είναι γεγονός ότι έχει επανέλθει ε, ο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ε, οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων λέγουν ε, ότι χρειάζεται προσοχή γιατί υπάρχουν κυβερνήσεις όπως αυτή του Κάμερον ε, που είναι πρόθυμοι να εθελοτυφλήσουν για να προωθήσουν τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα. Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά το τέλος ενός αιματηρού και βίαιου εμφυλίου πολέμου, τέσσερα χρόνια μετά τη γενοκτονία και τις σφαγές 70.000 ταμιλόφωνων, ε, στο τέλος του πολέμου. Ακόμα δεν υπάρχει ε, πλήρης, ε, διαφανής και αξιόπιστη διερεύνηση των εγκλημάτων της κυβέρνησης. Η ατιμορρησία κυριαρχεί ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανώτατους αξιωματικούς και για την κυβέρνηση. Βασικά θέλουν να ξεπλύνουν την κυβέρνηση για να βγει καθαρή από αυτή την υπόθεση. Ανεξάρτητη διεθνή έρευνα χρειάζεται εδώ και καιρό και θα πρέπει το συντομότερο να συσταθεί η Επιτροπή που να λογοδοτεί στα θύματα και τις οικογένειές τους. Η κοινότητα των ε, ομιλούν την ε, Ταμίλ ε, ήδη έχει αφαιθεί στη μοίρα της από τον ΟΗΕ. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να τους βοηθήσει, οργανώνονται σε ομάδες όπως η Ταμίλ Solidarity για την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Ευχαριστώ κύριε Μέρφη. Δέχεστε ερώτηση του συναδέλφου Ντίβα. Yes. Yes. ναι, παρακαλώ. Να ευχαριστώ κύριε Μέρφη. Καλωσύνη σας. Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μέρφη, αν μου επιτρέπετε, που είναι και εμπειρογνώμων ειδικό για την Σρι Λάγκα, να μου πει το εξή. Πόσοι Ταμίλ ζουν στη Σρι Λάγκα, πόσοι ζουν στο Νότο και πόσοι στο Βορρά. Και ποια ε, είναι ή ε, το ποσοστό του πληθυσμού των κατοίκων της πρωτεύουσας του Κολόμπο, οι οποίοι είναι Ταμίλ. Ευχαριστώ, κύριος Μέρφη. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Εγώ δεν βλέπω τον εαυτό μου, ε, δεν το θεωρώ εμπειρογνώμονα για τη Σιλάνκα. Θα ήθελα να έχω την ευκαιρία, όπως και εσείς, να πάω και επανειλημμένα η κυβέρνηση δεν μου δίνει βίζα. Γιατί έχω επικρίνει την καταστολή των Ταμίλ. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένους αριθμούς για το πόσοι είναι και πού ζουν. Προφανώς στο βορρά και στις βορειοανατολικές περιοχές, αλλά και στο Κολόμπο είναι πολύ και εκεί υφίστανται διακρίσεις. Και αν έκαθεν αυτό που λέω εγώ είμαι υπέρ μιας ενωμένης ε, μάχης και όσων ομιλούν ε, τη ε, γλώσσα άλλα και των Ταμίλ για δικαιοσύνη και ειρήνη στη Σιλάνκα. Λυπάμαι πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρο. δεν τον βλέπετε διμερό να τα πείτε. Ο κύριο Μπένιον, για 1,5 λεπτό. thank uh, thank you, you, Chair. Now Ευχαριστώ. Τώρα έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που τέλειωσε η σύραξη μεταξύ των τρικών του Νταμίλ και τη ε, κυβέρνηση, και εξακολουθούν να υπάρχουν καταγγελίε από ομάδε ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι συνεχίζεται η τιμωρησία ε, για όσου έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα και εγκλήματα πολέμου. όμω το σημερινό ψήφισμα είναι ισορροπημένο και αναγνωρίζει και την πρόοδο που έγινε κυρίω ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση, την αφαίρεση των αρκών και τι ε, επιτυχείς δημοτικές εκλογές που είδαμε ε, στο Βορρά όμως θα πρέπει ε, να γνωρίζουν οι άνθρωποι τι έγινε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στους συμπολίτε τους και μια ανεξάρτητη έρευνα για τις παραβιάσεις ε, του διεθνούς δικαίου που έγινε και από τις δύο πλευρές, το προλαμβάνω και από τις δύο πλευρές της σύραξη αυτή είναι απολύτως απαραίτητη και επιγόντες και θέλουμε να καλέσουμε την κυβέρνηση Σρι να προβεί σε μια ανεξάρτητη έρευνα το συντομότερο. Αν η κυβέρνηση δεν ε, ξεκινήσει μέχρι το Μάρτιο 2014 μια αξιόπιστη διαδικασία, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ξεκινήσουν μια δική του ανεξαρτητή έρευνα. Επομένω, ε, καλό δεν είπα αρμοστή του ΙΕ τώρα προδραστικά να ξεκινήσει επαφές με την κυβέρνηση για ένα τέτοιο αποτέλεσμα και ε, θα ήθελα να υπάρξει αυτή η ε, έναρξη της ε, έρευνας στην ίδια βάση όπως η έρευνα που γίνεται για τους εξαφανισμένους, για τους αγνοούμενους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπένιον. Επιτρέπετε διάμεση ερώτηση του κυρίου Λάινεν. Έχει ερώτηση ο κύριος Λάινεν, τον αφήνετε να την κάνει. Ναι. <laughs> Είναι από την αριστερή πλευρά, μην κοιτάτε από εκεί. Ε, μετά από 30 χρόνια εμφυλίου πολέμου ήταν μεγάλο το χάος στη Σρι Λάνκα. Ε, Λέγουν ε, ορισμένοι ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, όχι αρκετά. Μιλάτε για ισόρροπο ψήφισμα και ζητάτε μια ε, συνολική διερεύνηση μέχρι το Μάρτιο του 2014, μέσα σε τρεις μήνες. Σας φαίνεται ρεαλιστικό αυτό ε, το τελεσίγραφο. Με δικά σας λόγια, ίδιος είπατε ότι είναι το χρόνο, αλλά το Μάρτιο του 2014 είναι τελείως ανεδαφική αυτή η προθεσμία. Ευχαριστώ. Well, certainly. Ναι, βεβαίω συμφωνώ ότι δεν θα ήταν ρεαλιστικό να ολοκληρωθεί μια έρευνα μέχρι το Μάρτιο του 2014, αλλά απλώ ζητάμε να ξεκινήσει η έρευνα αυτή. Και το χρονοδιάγραμμα σχετίζεται με τις συνεδριάσεις του ΙΕ το Μάρτιο του 2014. Ζητάμε λοιπόν απλώ να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία μέχρι τότε και η διαδικασία της έναρξης ε, Απλώς περιλαμβάνει το εξή να στείλει ο Πρόεδρος ε, την κοινοποίηση και να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη προκειμένου να σχηματιστεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Μπένιον. Τελευταίος από τους συντάκτες των ψηφισμάτων ο κύριος Λίζεκ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπα, αυτοί συνάδελφοι, είναι πολύ καλό που συζητάμε την κατάσταση στη Σρι Λάγκα για μια ακόμη φορά. Ξέρουμε ότι πέρασε τεράστια δεινά η χώρα αυτή, πολλές χώρες, πολέμα, εγκλήματα, οιασμοί, δολοφονίες, ε, επικισμοί κτλ. Θα μπορούσαμε να συντάξουμε ένα μακροσκελέστατο κατάλογο. Ευτυχώς ε, για τέσσερα χρόνια τώρα υπάρχει ειρήνη στην περιοχή. Βέβαια, ε, θα πρέπει να νοικοδομηθούν οι κρατικές δομές. Και μπορούν να βοηθήσουν ευρωπαϊκές χώρες όπως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει ε, μακρά ιστορία στη σχέση του με τη χώρα αυτή. Θα μπορούσε να γίνει μεταφορά τεχνογνωσίας για παράδειγμα για να νοικοδομηθούν οι κρατικές δομές. Και ελπίζουμε η χώρα αυτή να ευημερήσει σε συνθήκες ειρήνης και οι διαφορετικές αθλητικές ομάδες να μπορέσουν να συνεπάρχουν ειρηνικά. Σίγουρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται έρευνα. Ελπίζω να μπορέσουν να τα λύσουν μόνοι τους ε, στη Σριλάνκα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Λίζε. Εδώ ολοκληρώνονται λοιπόν οι συντάκτες και εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Πρώτος ο κύριος Πόσελτ από το ΕΛΚ ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, στη Σιλάνκα πρόκειται για εθνοτική σύραξη. Ε, σε μία μεταπικιακή κατάσταση γεννήθηκε. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος που έκαναν παλιές απικιακές δυνάμεις ίσως, αλλά να προσπαθήσουμε από την κατάπαυση του πυρός ή το μη πόλεμο, να μεταβούμε σε μια πραγματική γνήσια ειρήνη. Για να γίνει αυτή θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη και πραγματική ειρήνη γίνεται μόνο όταν υπάρχει εσωτερική ειρήνη. Οπότε, από τη μια να δίνουμε τα δικαιώματα σημαντικό για πλειονότητες και μειονότητες, αλλά και το εσωτερικό ε, ε, ειδικό βάρος έχει σημασία και οι σχέσεις και ε, για μένα η ημερομηνία είναι επίσης σημαντική. Δεν τρέφονται αυτά πάτες ότι θα έχουν λυθεί τα πάντα, αλλά εάν το αναβάλουμε θα το αναβάλουμε για το Αγίου ποτέ, όπως βλέπουμε να γίνεται σήμερα στη Σερβία και αλλού. Αυτά τα εγκλήματα χρειάζονται επεξεργασία και είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Και απευθύνω έκκληση στην πλειοψηφία αυτό να το κατανοήσει, να το αναγνωρίσει. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ, η κυρία Γκέριγκερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Το Νοέμβριο ε, φιλοξένησε τη συνέντευξη τη κοινοπολιτεία Σρι Λάγκα. Υπάρχουν κριτικέ ε, από την εθνική κοινότητα, ε, ότι δηλαδή δεν έχουν προσαρθεί από τις δικαιοσύνη, οι υπεύθυνοι αυτή τη σύγκρουση, που κρατούσε 26 χρόνια με πάρα πολλού νεκρού, εκτοπιστέντε κτλ. Το θέμα είναι σίγουρα να εξομαλυνθεί η χώρα, το βόρειο τμήμα, να κλείσουν οι καταβλισμοί των προσφύγων και να ε, καθαρίσει από τις νάρκες ε, η περιοχή για να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν εκεί οι κάτοικοι. Ξέρουμε ότι πριν τα τέλη του εμφυλίου πολέμου το 2009 έγιναν διάφορα ε, έκτροπα και κλίματα. Έχει τα στοιχεία στα χέρια του. Δύσκολο είναι το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών μετά από τόσα χρόνια εμφυλίου πολέμου, αλλά χρειάζεται για την συμφιλίωση και τη δημοκρατία κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέρινγκερ. Για ένα λεπτό, ο κύριος ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Οι πολίτες της Τριλάνκα έχουν υποφέρει πολλά χρόνια ε, τρόμου από τους ε, τα μήλα. Μέχρι βέβαια και ο στρατός έκανε ε, εγκλήματα, χρησιμοποίησαν ε, ματηριδία και οι δύο πλευρές σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΑ. Θα πρέπει να γίνουν λοιπόν οι προσπάθειες της επανασυμφιλίωσης όλων των πολιτών από όλες τις αθλητικές ομάδες και απευθύνω έκκληση στην κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων. Η αποκέντρωση είναι η βάση. Οι ομάδε θα μπορέσουν έτσι να ελέγχουν την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα σε ένα επανενωμένο κράτο. Επίση, είναι απαραίτητο να διαλευκανθούν, να επιληθούν ε, οι υποθέσει, ε, τα εγκλήματα. Θα πρέπει να ε, τιμωρηθούν οι ένοχοι. Ξέρουμε ότι υπάρχει ακόμη ε, διαφθορά, υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι, συνεχίζονται τα εγκλήματα. Πρέπει να βοηθήσουμε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Σρι Λάγκα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ αυτό το ψήφισμα δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων στη Σιλάκα. Για να πιστεί κανείς, ε, αρκεί να διαβάσει τι λέει ε, ε, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Είναι όλο και πιο αυταρχική η κυβέρνηση της χώρας. Οι ΜΚΟ καταγγέλουν ναι, επιδείνωση της καταστολής στη χώρα αυτή που αφορά κυρίως τα ΜΙΛ. Δεδομένης κατάστασης αυτής λοιπόν, πώς να αποδεχτεί κανείς ότι αυτοί που ζητούν στην Ευρώπη καταφύγιο ε, ε, ε, τους θέλουν πίσω στο Κολόμπο με κίνδυνο χάσουν τη ζωή τους. Έχω στη μνήμη μου ένα νέο 30 ετών, Χάντζεν Βαν. Ήταν πρόσφυγας εδώ στο Στρασβούργο ακριβώ. και τον επαναπάτρισαν στη Στριλάνκα παρά την κινητοποίηση κατά της έκδοσης. Έξι μήνες μετά έχασε τη ζωή του γαζωμένος από σφαίρες. Ε, ο θείος του ε, επίσης ε, βασανίστηκε. αυτά όλα είναι αφόρητα. Τέτοια δράματα δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Βερζιά. Ο κύριος Δίβα έχει ερώτηση, επιτρέπετε. Πείτε, Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς. Ναι, κυρία Βερζιά, γνωρίζει κυρία Βερζιά Πρόεδρε ότι το Κολόμπο, η πρωτεύουσα της Σρι Λάγκα, όπου είναι μια πόλη μειονοτική με 64% του πληθυσμού να ε, ομιλούν ταμίλ και όχι, ε, και όχι σριλανκέζικα. Περί τίνος πρόκειται, μα γιατί πράγμα μιλάει. Η κυρία Βερζιά, ζητώ συγγνώμη. Και το πρόβλημά σας ποιο είναι. Το θέμα δεν είναι ποιος μιλάει σε, ε, ε, Σριλανκέζικα και ποιος μιλάει Ταμίλ. Το θέμα είναι να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, επιδεινώνεται. Υπήρχε μια μηδρή ελπίδα συμφιλίωσης, έχει παρέλθει και θα πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως λέει ο ΟΗΕ. Και εμείς υποστηρίζουμε την ύπατη αρμοστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Και τώρα ο συνάδελφος Μάγερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 26 χρόνια ε, εμφύλιος πόλεμος με σοβαρές ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σύμβαση της Γενέβης, Εκατέρωθαν. Από το 2009 λέει η κατάσταση είναι σταθερή, de facto ε, κυριαρχία του αποσχιστικού βορρά έχει τερματιστεί. Ανθρώπινα δικαιώματα γίνεται λόγος για 30.000 ε, μεταξύ αυτών πολλοί δημοσιογράφοι νεκροί αγνοούμενοι. Μέχρι και 80.000 ακούμε ε, πρόσφυγες από το Βορρά λόγω του εμφυλίου που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις συστήσεις τους. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καλέσει την κυβέρνηση να τα διευκρινίσει αυτά, ε, να σταματήσει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα το κάνει αυτό η Ένωση, αλλά είναι πολύ πιο απλό να χτυπάμε το χέρι μας στο τραπέζι απέναντι σε χώρες όπως η Σρι Λάγκα παρά η μεγάλη χώρα, η Κίνα ας πούμε. Θα πάω στη Σρι Λάγκα να δω τη χώρα, είμαι πολύ αισιόδοξο για το μέλλον της, θέλω η διεισόμαση να διαπιστώσω τι συμβαίνει εκεί. Ευχαριστώ κύριε Μάιερ. Ο κύριος Δίβα για δύο λεπτά. Ε, Mr. thank Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρέπει να δηλώσω συμφέρον, προφανές. Γεννήθηκα στη Σρι Λάγκα, ο παππούς μου ήταν γερουσιαστής και ιδρυτικό μέλος του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης. Είναι αξιοθρύνητα ε, αυτά που συνέβησαν. 60.000 ζωές οι τρομοκράτες που εξεγέρθηκαν ε, ε, προκάλεσαν. Είναι κρίμα που το έχει ξεχάσει το κοινοβούλιο αυτό και ε, συνεχίζει με διεθνείς ε, κρίσεις για το πώς τέλειωσε ο πόλεμος. 30 χρόνια οι κρατικοί παράγοντες υπερασπίζονταν το κράτος δικαίου απέναντι σε μη κρατικούς παράγοντες που τρομοκρατούσαν ε, ε, αθώους πολίτες και τους χρησιμοποιούσαν ως ανθρώπινες ασπίδες. Έχει ιστορία 2.600 ετών η Σιλάνκα υπερήφανη και ενωμένη. 14 φορές υπέστη εισβολή από ένα δυνάμεις από την Υπηρωτική Ινδία και 14 φορές οι ε, βασιλείς της την απέκρουσαν. Η Σρι Λάνκα είναι και η πιο ευρωπαϊκή εντό εισαγωγικών από οποιαδήποτε άλλη ασιατική χώρα. Έχει 500 έτη ε, ε, ευρωπαϊκής ιστορίας και πολιτισμού. Πρώτα ήταν οι Πορτογάλοι, μετά οι Ολλανδοί, μετά οι Άγγλοι. Το 1928 ήταν δημοκρατική χώρα πολύ πιο από τα 19 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα θεωρούν απολύτω θεμητό να δίνουν μαθήματα δημοκρατίας. Όλα αυτά είναι ε, ε, ε, για γέλια. Αυτά που είναι για γέλια όμως γίνονται γελία όταν βγάζουμε εδώ πέρα στο κοινοβούλιο τελεσίγραφα ότι θα πρέπει να κάνει χώρα αυτό το τάδε ή το δίνα μέχρι την τάδε ή τη δίνα ημερομηνία ε, ε, με κυρώσει ε, να επαπειλούνται. Τι είμαστε στην εποχή των απικιών, είναι τελείως αντιπαραγωγικά αυτά και κάνει την κυβέρνηση της χώρας σήμερα ακόμα πιο δημοφιλή. Θα πρέπει να οικοδομήσουμε ανταυτού η ειρήνη βιώσιμη και διαρκή. Ευχαριστώ κύριε να οικοδομησουμε ανταυτου κύριε Πρόεδρος διακόπτη τον ομιλητή. Κύριε Ντίβα, επιτρέπετε ερώτηση του κυρίου Μέρφυ. Επιτρέπετε την ερώτηση του κυρίου Μέρφυ. Uh, Ευχαριστώ που δεχτήκατε την ερώτηση. Πρόσεξα ότι κάνατε μια διάκριση μεταξύ τη ε, κρατική βία και τη μη κρατική βία. Κατά την άποψή του είναι αποδεκτό το κράτο, να προσβαίνει σε σφαγιασμό ανθρώπων ε, και να ε, έχει εξαφανίσει ανθρώπου και να καταστήλει τα μέσα με 60 μέρε, επειδή απλώ είναι το κράτο, Δηλαδή κατηγορούμε λιγότερο το κράτο από ότι άλλου όταν αυτοί εμπλέκονται σε βιοπραγίε απάντηση. Αν μου άκουσε σωστά ο κύριος Μερφή... Ε, αν με είχε ακούσει σωστά, θα καταλάβαινε ότι εγώ δεν δικαιολόγησα την κρατηδία. Ε, είπα, ε, μίλησα για υπεράσπιση του κράτους δικαίου για 30 χρόνια. Οι κρατικοί παράγοντες υπεράσπισαν το κράτος δικαίου και αν δείτε πώς έγινε ο πόλεμος για 30 χρόνια, ο Νότος έτρεφε το Βορρά, τον πληθυσμό που έβαζε βόμβες και έστελνε τρόφιμα εκεί πάνω. Εδώ μιλάμε για τρομοκρατικές πράξεις από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που δεν έχει καμία σχέση με τον πληθυσμό των Ταμίλ. Και διακόπτει ο πρόεδρος τον ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντίβα. Ερχόμαστε στο Catch the Eye και σας παρακαλώ να κατανοήσετε ότι θα δώσω το λόγο σε πολύ λίγους όσους δεν μίλησαν ακόμα. Ο κύριος Κίνερ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Oh, Λειτουργεί μάλιστα. Θα προσπαθήσω να μην ε, μακρηγορήσω πάρα πολύ. Απλώς να πω ότι το ψήφισμα αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο και έγκαιρο. Η πρόοδος στη Σιλάνκα ήταν αργή και σε πάρα πολλούς ε, περιοχές ε, και τομείς ε, πρέπει το καθεστώς να οικοδομήσει τη φήμη του και να αντικρούσει ε, τους ισχυρισμού για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο παρελθόν και σήμερα. Αρκεί να δείτε το έργο της Ναβι Πίλη από τα Ηνωμένα Έθνη για να δείτε ότι υπάρχουν κάποια κρεμή ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Κάποια αυτά τα θέματα εξακολουθούν ε, να σχετίζονται με εκατοντάδες χιλιάδες, χιλιάδες εξαφανισμένους ε, και με τη δολοφονία ανθρώπων ανθρώπων που εργάζονταν στην παροχή ανθρωπιστική βοήθεια. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε να κάνει τίποτα γι' αυτά και αν ε, δεν υπάρχει πίεση από τα μέσα και από τα έξω, από ό,τι φαίνεται και πάλι δεν θα σημειωθεί κάποια πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκίνερ. Τελευταίος, συνάδελφος Ρέπο για το κατσί. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, σίγουρα εκτιμώ όλο ιδιαίτερο την εμπειρία του κύριου Ντιβάν. Κατάλαβα καλά τα προβλήματα τη Λάγκα χρονολογούνται από την εποχή του εμφύλιου πολέμου που τερματίστηκε το 2009. Πρόκειται για ε, φρικαλές ε, βιαιότητες, ε, δεκάδες χιλιάδες ε, ε, θύματα μέχρι και σε νοσοκομεία, επιθέσεις κτλ. Ο ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ που επισκέφθηκε την περιοχή έκανε δηλώσεις και πρέπει να τι λάβουμε υπόψη. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, δραστήριοι σε ό,τι αφορά την επανασυμφιλίωση. Σίγουρα δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα εγκλήματα πολέμου. Τα φαινόμενα ατιμορρησία πρέπει να πάψουν. Ακούμε ότι κάτι, μάλλον έχουν ε, πει πολλά πράγματα κάτι και στη Σρι έχουμε ακούσει διάφορες ιστορίες. Η Σρι θέλει να έχει διάλογο με την εθνική κοινότητα, αλλά με ανησυχούν πάρα πολύ τα στοιχεία που μιλούν για επιθέσεις ε, κατά εκκλησιών ε, και μουσουλμανικών τεμενών. Πρέπει να υπάρχει θρησκευτική ελευθερία. Ευχαριστώ. Κύριε Ρέπο, ολοκληρώνεται η διαδικασία Κατσέη. Και για να κλείσει η συζήτηση το λόγο έχει ο Επίτροπο κ. Τσόλο. Ευχαριστώ. Χαιρετίζουμε την υιοθέτηση ενό ε, ψηφίσματο εκτάκτη ανάγκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατία και την κατάσταση του δικαίου στη Σιλάνκα. Όπω αναφέρεται στο ψήφισμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει επίση ότι η Σιλάνκα με τη βοήθεια τη διεθνού ε, κοινότητα ε, έχει προβεί σε σημαντικέ βελτιώσει από το τέλο τη σύρεξη, κυρίω σε ό,τι αφορά την αφαίρεση των ερκών και την αποκατάσταση των υποδομών. Επίση, Επίσης χαιρετίζουμε τις πρώτες εκλογές του Επαρχικού Συμβουλίου του Βορρά και Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια ε, ουσιαστική συνεργασία μεταξύ αυτού του Συμβουλίου και της κεντρικής κυβέρνησης. Όμως ε, και άλλες προκλήσεις παραμένουν να αντιμετωπιστούν στη Σρι κυρίως ότι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις θρησκευτικέ ε, ελευθερίες και ατομικές ελευθερίες, την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και του κράτους δικαίου. Επίσης πρέπει να αναλυφθεί πλήρης ευθύνη για τα εγκλήματα του παρελθόντος. Έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε θερμά την κυβέρνηση της Σρι να λάβει πρόσθετα μέτρα για να θέσει σε εφαρμογή τι συστάσει ε, που διατυπώθηκαν από τη δική της Επιτροπή Διδαγμάτων και Συμφιλίωσης και να κάνει μια εξάρτητη έρευνα για τις υποτιθέμενες περιβιάσεις του διεθνού δικαίου τέτοιες εκκλήσεις έγινε και από άλλους διεθνείς εταίρους ε, και η πρόοδος θα αξιολογηθεί πριν το επόμενο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Μάρτιο του 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ στη διαδικασία. Εμεί, προ την κατεύθυνση αυτή σημειώσαμε ε, με ικανοποίηση την σύσταση μια επιτροπής για την διερεύνηση τη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Σρι Χαιρετίζουμε την επίσκεψη τους είπα το Ερμοστή των Ηνωμένων Εθνών ε, και το Αξιωματούχου των Ηνωμένων Εθνών για τους εκτοπισμένους ε, και ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση να ε, διευκολύνει την επίσκεψη των αξιωματούχων του ΟΗΕ στη χώρα αλλά και της ομάδας εργασίας για τις εξαφανίσεις για τους αγνοούμενους. Επίσης ενθαρρύνουμε τη Σιλάνκα να ενταχθεί σε ένα διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλους διεθνείς εταίρους ε, που ίσως μπορέσουν να συνεισφέρουν για τι ε, δύσκολες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπιστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προσφέρει την υποστήριξή τη στην κυβέρνηση της Σρι για να τη βοηθήσει να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις και να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους πολίτες. Της ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσόλος. Έχουν κατατεθεί έξι ψηφίσματα συνολικά για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, η οποία και ολοκληρώνεται και περνούμε μέσω στι ψηφοφορίε. Αρχίζουμε με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Πέντε πολιτικές ομάδες έχουν καταθέσει ψήφισμα. Ε, τροπολογία 1 υπέρ. Κατά